με πολύ, σημαντικές, ε, με πολύ σημαντικό αντίκτυπο για τη σταθεροποίηση του ευρώ αλλά και τη εσωτερικής Αγόρα. Ευχαριστώ. Είχαμε μία πρόταση ψηφίσματος για την περάτωση αυτής της συζήτηση. Η συζήτηση έληξε. Η ψηφοφορία θα δεξαχθεί αύριο στις 12 το μεσημέρι. Το επόμενο σημείο στη στη διάταξη είναι η έκθεση του κυρίου David Μάρτιν, εξαίρεση ορισμένων χωρών από τον κατάλογο των περιφερειών ή των κρατών που έχουν ολοκληρώσει διαπραγματεύσει. Το λόγο έχει ο εισηγητής, ο κύριος David Martin, συνάδελφος κύριος Μάρτιν, για τέσσερα λεπτά. Thank you very much, President. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει καθεστώς προτιμησιακό σε κράτη της ε, Αφρικής Καραϊβικής και του Ειρηνικού με μια εξαίρεση στο το 2006, μια παρέκκληση δηλαδή από τον ε, Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου που μας επέτρεπε να δώσουμε αυτές τις μονομερείς συμφωνίες, ε, τις προτιμήσεις δηλαδή, η οποία όμως θα έπρεπε να εκπνεύσει με την υπογραφή των ΣΟΕΣ, δηλαδή των Συμφωνιών Οικονομικής εταιρική Σχέσης, που όμως δεν πραγματοποιήθηκε και έτσι από την απόφαση του 2007 χρειάστηκε να δοθεί μία λύση μετάβαση με αδασμολόγητες και χωρίς ποσοστώσεις δυνατότητε πρόσβασης στις αγορές για τις χώρες αυτές οι οποίε έχουν μόνο γράψει αλλά δεν έχουν ακόμα ε, υπογράψει ή επικυρώσει τι συμφωνίε αυτέ. Θεωρεί λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι αυτή η προσωρινή λίστα πρέπει να ε, τερματιστεί η πρόταση της ΔΕ είναι αυτή η προτιμησιακή ε, μεταχείριση να λήξει από 1η Ιανουαρίου του 2014. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Πρόεδρε, κατά την άποψή μου, δεν έχει απόλυτο δίκιο, μόνο κατά το ίμιση. Είναι βεβαίω ήταν προσωρινή λύση αυτή η συμφωνία ε, και όντω θα πρέπει να έρθει το τέλος της κάποια στιγμή. Από την άλλη όμως οι αναπτυσσόμενες χώρες εκτός των κρατών ΑΚΕ που βλέπουν ότι οι χώρες σε επίπεδο αντίστοιχο οικονομικό με το δικό τους έχουν πλεονεκτήματα που ε, οι ίδιες δεν γνωρίζουν. Και σε αυτό έχει δίκιο η Επιτροπή. Αλλά θα πρέπει όλα αυτά να τα δούμε και μέσα στα τρέχοντα πλαίσια των ε, τρεχουσών συμφωνιών οικονομική εταιρική σχέση και να μην δημιουργήσουμε την εντύπωση, το φόβο ή όπω αλλιώ θέλετε πείτε το, ότι εκφοβίζουμε τις αφρικανικές χώρες ε, έτσι ώστε αυτές να υπογράψουν ε, ή να κυρώσουν τις συμφωνίες οικονομικής εμπορικής σχέσεως και δεν τους δίνουμε περιθώριο οικονομικό. Γι' αυτό λοιπόν θα πρότεινα να μετακινηθεί η προθεσμία από την 1η Ιανουαρίου 2014 στην 1η Ιανουαρίου 2016 έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα να δουν οι χώρες αυτές του ΑΚΕ ότι όντως ε, τελειώνουν, τερματίζονται αυτέ οι προτιμησιακέ σχέσει, αλλά ταυτόχρονα θα έχουν και ένα περιθώριο για ανάπτυξη των διαπραγματεύσεων. Κάποιοι συνάδελφοι ξέρω ότι θα πούν, όπω μου έχουν ήδη πει, ότι αποτελεί μια παραπέρα παράταση τη προθεσμία. Όχι, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν είχαμε μέχρι τώρα προθεσμία. Πρόκειται για μια πρώτη πρόταση για προθεσμία, αυτή που συζητούμε τώρα. Και εάν εγκριθεί, θα είναι σαν γραμμένη, σε σε μάρμαρο, δεν θα δοθεί δηλαδή περαιτέρω περιθώριο, περιθώριο προθεσμία ούτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και, πάση περιπτώσει, δεν θα μπορεί να δοθεί χωρί συμφωνία Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και άλλωστε αμφισβητώ και αν θα είναι διατεθειμένη η Επιτροπή να προσφέρει άλλη λύση μεταγενέστερη. Ε, δίνεται η εντύπωση από την επιχειρηματολογία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι η πρώτη Ιανουαρίου του 2014 θα δώσει περισσότερο κύρος στις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης εάν τηρηθεί αλλά όπως και άλλοι συνάδελφοι εγώ θεωρώ ότι αυτό δεν ισχύει γιατί οι περισσότεροι θεωρούν ότι δεν είναι λογικός αυτός ο στόχος ε, του 2014 και αν εγκρίνουμε το 2014 φοβόμαι ότι θα, εγκρίνω, αποκλείσουμε από το πλαίσιο αυτό, από το σύστημα αυτό 17 χώρες ενώ με το 2016 μπορεί να, μπορούμε να ορίσουμε και αυστηρό στόχο αλλά και ευκταίο στόχο, εφικτό στόχο. Έτσι λοιπόν για λόγους τόσο λογικής όσο και λόγους οικονομικής σκοπιμότητας θεωρώ το 2016 είναι στόχος εφικτός, είναι στόχος που μπορούμε να τηρήσουμε και ελπίζω ότι θα μπορέσω να πείσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αλλάξει το στόχο. Έτσι η Επιτροπή θα έχει και έναν αυστηρό στόχο μια ε, αίρεση ε, για την λήξη των συμφωνιών, αλλά και θα δώσει ένα περιθώριο στις χώρες αυτές. Ευχαριστώ πολύ και τώρα θα παρακαλούσα τον Επίτροπο De να λάβει το λόγο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Uh, uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του Κοινοβουλίου. Ορισμένοι από εσά πήρατε μηνύματα κατεπήγοντα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχίσει να βοηθά τις αναπτυσσόμενες χώρες η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το οποίο δεν σας είπαν όμως είναι το εξή. Μέχρι το τέλος του 1990 εμείς δίναμε στις χώρες ΑΚΕ ειδικέ μονομερείς δασμολογικές ρυθμίσεις πέρα από τις συμφωνίες που είχαμε κάνει για τις εμπορικές προτιμήσεις με άλλες χώρες σε σχέση με τις συμφωνίες της Γενέβης. Τώρα πλέον δεν μπορούμε να κάνουμε διακρίσεις ανάμεσα σε χώρες που βρίσκονται στην ίδια οικονομική κατάσταση. Μόνο με μία ρύθμιση την οποία είχαμε κάνει για τελευταία φορά μέχρι το 2007. Εν τω μεταξύ πιστεύαμε ότι θα έπρεπε να έρθουμε στο επίπεδο που προβλέπει ο ΠΟΕ. Το 2000 είχαμε υπογράψει συμφωνία Κοτονού με τις χώρες ΑΚΕ είχαν συμφωνήσει να εξυγχρονίσουν τις εμπορικές τους σχέσεις. Να μην ξεχνάμε ότι μέχρι τότε ακόμα και αυτές οι πολύ γενναίες προτιμήσεις δεν είχαν βελτιώσει τις εξαγωγές ΑΚΕ προς την Ευρώπη. Από το 67 μέχρι το 99 το ποσοστό των χωρών ΑΚΕ στις εισαγωγές πήγε από 7,7 σε 8,7. Δηλαδή συμφωνήσαμε στο Κοτονού στα πλαίσια του άρθρου 16 της συνθήκης να συνάψουμε μια νέα εμπορική συμφωνία η οποία να είναι συμβατή με τον ΠΟΕ. Ήταν μια πρόταση που είχε οικονομικό νόημα λόγω ακριβώς των παλιών εμπειριών που ήταν αρνητικές με τη χρήση των εμπορικών προτιμήσεων. Ήταν και κάτι που ήταν συμβατό με την πολιτική ατμόσφαιρα εκείνη τη εποχή. Η διεθνής κοινότητα είχε κατανοήσει ότι οι αναπτυξιακές πολιτικές δεν στηρίζουν τις χρηστές πολιτικές. Η εμπορική πολιτική έπρεπε να αντικατοπτρίζει αυτή την αντίληψη και το έχω πει στο παρελθόν και θα το ξαναπώ. Η πολιτική αξία των διμερών εμπορικών σχέσεων <coughs> είναι ότι δίνουν τη δυνατότητα στους θεσμούς να διαχειριστούν τις ανηλυμένες εμπορικές υποχρεώσεις. Πέρα από τα κίνητρα προς δύο κατευθύνσεις των εμπορικών συναλλαγών, οι ρυθμίσεις αυτές οι ε, δασμολογικές επιτρέπουν επίσης και ε, βήματα προόδου στον τομέα της διαφθοράς. Τι άλλο θέλω να πω. Το 2007 μόλις είχαμε κλείσει τις διαπραγματεύσεις είπα με τις μισές από τις χώρες ΑΚΕ η Ευρωπαϊκή Ένωση με καλή πίστη πέρασε ένα νόμο ο οποίος επέτρεπε στους εταίρους μας τους εμπορικούς να ε, εξάγουν τα προϊόντα τους χωρίς ε, επιβολή ποσοστώσεων και χωρίς την επιβολή δασμών. Λέγοντας όμως ότι οι εταίροι μας μέχρι το 2000 ε, μετά από δύο χρόνια θα είχαν εξυγχρονίσει τους μηχανισμούς με τους οποίους συμμετείχαν στις εμπορικές συναλλαγές. Οι περισσότερες χώρες το έκαναν αυτό. 18 χώρες μέχρι το τελευταίο χρόνο δεν το είχαν κάνει εννέα χώρες που έχουν μείνει είναι λιγότερο αναπτυγμένες και συνεχίζουν να έχουν ε, εμπορικές προτιμήσεις γιατί δεν είναι σε θέση να συμμετέχουν σε άλλες διαδικασίες και αυτές οι χώρες επηρεάζονται από τις ε, χώρες που μιλάμε, από τις ε, ρυθμίσεις που μιλάμε σήμερα. Μποτσουάνα, Καμερούν, ε, Ακτή ελεφαντόδοντος, Σουαζιλάνδη και Μποτσουάνα. Έχουμε προχωρήσει λοιπόν. Βλέπουμε ότι άνω των 80 χωρών είχαν το 2011 μέσα σε τρία χρόνια κάνει τις ρυθμίσεις οι οποίες χρειαζόντουσαν. Η εικόνα η γενικότερη είναι κάτι το οποίο μας κάνει θα έλεγα υπερήφανους. Συνεχίζουμε τις διαπραγματεύσεις στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας είπα και νομίζω ότι υπάρχουν λίγες εκκρεμότητες με την κοινότητα της Ανατολικής Αφρικής, με τη Δυτική Αφρική και με τους εταίρους μας είπα στα πλαίσια της αναπτυξιακής κοινότητας του νοτιού τμήματος της Αφρικής ΑΔΕΚ. Έχουμε προχωρήσει στις ε, διαπραγματεύσεις με την Καραϊβική με την Παπούα Νέα Γουινέα και με τις υπόλοιπες χώρες. Κάποιες από τις χώρες αυτές συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις έτσι ώστε να προχωρήσουν σε ολοκληρωμένες περιφερειακές συμφωνίες. Τι, περιοχ... τι περιέχει η συμφωνία αυτή. Βασικά η συμφωνία αυτή καλύπτει τα προβλήματα του παρελθόντος. Είχαμε ξεκινήσει από το 2007 Δεν μιλάμε εμείς αυτή τη στιγμή για τις ε, συμφωνίες ΕΠΑ οικονομικής εταιρικής σχέσης, αλλά είναι συμφωνίες που καλύπτουν όπως είπα τα κενά του παρελθόντος και δεν στρέφονται στο μέλλον. Αυτοί που θέλουν την παράταση του status quo ε, θα έλεγα ε, αντιστέκονται αλλά διαρωτώ με μήπως εμείς θα πρέπει να ακολουθήσουμε δεν κάναμε τις προσπάθειες που έπρεπε από το 2004 και μετά. Γιατί θα πρέπει ένας επιχειρηματίας από την Αμίμπια ή από την ακτή του Ελεφαντοστού να μην μπορεί να και... και που εξακολουθεί και έχει ανάγκη και προμηθεύεται ευρωπαϊκά μηχανήματα σαν παράδειγμα να πληρώνει πάρα πολύ υψηλούς δασμούς γι' αυτό. Πόσες νέες θέσεις εργασίας θα μπορούσαν να δημιουργηθούν με την κατάργηση των δασμολογικών επιβαρύνσεων. Γιατί θεωρούμε τις χώρες αυτές ικανές να εξάγουν μόνο βασικά προϊόντα ανεπεξέργαστα. Είμαστε μακριά από τη σημερινή πραγματικότητα. Ε, πολλές φορές θέλουμε να κάνουμε το καλό και δεν το κάνουμε ή κάνουμε κάτι το οποίο δεν αρκεί. Ε, τον Φεβρουάριο του 2010 είχα αναλάβει την υποχρέωση κύριε Πρόεδρε να ενισχύσω ακόμα περισσότερο ε, το σύστημα αυτό. Εκείνη την εποχή είχα εκφράσει και τη φιλοδοξία μου να προχωρήσουμε με τις συμφωνίες ΕΠΑ έτσι ώστε να καταστούν συμβατές με τις ρυθμίσεις του ΠΟΕ. Σαν Επίτροπος είμαι φυσικά δεσμευμένος από τον κοινοτικό νόμο. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και λόγω των πεπιθήσεων ότι η χρήση του ελευθέρου εμπορίου βοηθά όλες τις χώρες, θα συνεχίσω να υποστηρίζω την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να τροπολογηθεί ο κανονισμός με, από το 2014 ε, και μετά. Ελπίζω να σας πείσουμε γι' αυτό. Επίτροπε, τώρα περνάμε στους ομιλητές εξ ε, των πολιτικών ομάδων. Ο κύριος Φιέλνερ από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Αν έχει νόημα αυτή η συζήτηση, θα πρέπει να αρχίσουμε από την αρχή. Να δούμε δηλαδή ποιος είναι ο λόγος για όλα αυτά. Γιατί δηλαδή οι παλές εμπορικές συμφωνίες με τις Δυτικές Ινδίες ή στον Ειρηνικό θεωρούνται ε, μη βάσιμες. Γιατί γίνονται διακρίσεις, γιατί θεωρείται ότι γίνονται διακρίσεις και γιατί θα πρέπει να κινηθούμε σε αυτές τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης. <clears throat> Πέρασε πολλής χρόνος και θα πρέπει να φτάσουμε σε αυτές τις ε, συμφωνίες το ταχύτερο δυνατόν γιατί έτσι θα γίνουν οι σωστές επενδύσεις και θα υπάρξει και καλύτερη διακυβέρνηση σε αυτές τις χώρες. Ο μόνος λόγος για τον οποίο υπάρχουν αυτές οι προτιμησιακές εμπορικές σχέσεις είναι για να καλύψουμε το χάσμα μεταξύ των παλαιών παράνομων συμφωνιών και των νέων. Ήταν αρκετά αυθαίρετες και το όλο ζήτημα είναι πόσος καιρός θα χρειαστεί μέχρι ώστε να αρθούν αυτές οι αφαίρετες συμφωνίες. Άλλοι λένε 2016, 2017. Άλλοι δεν μπορούν να το προσδιορίσουν. Εν πάση περιπτώσει είναι γεγονός ότι έχουν περάσει 12 χρόνια και νομίζω ότι αδικήσαμε και άλλες φτωχές χώρες εκτός ΑΚΕ. Και γι' αυτό θα πρέπει να αναθεωρήσουμε την πολιτική μας. Γι' αυτό θα πρέπει να ορίσουμε μια προθεσμία για τη θέση σε ισχύ αυτών των συμφωνιών. Θα πρέπει να είμαστε δίκαιοι γιατί οι ΣΟΕΣ αυτές, οι Συμφωνίες Οικονομικής και Εταιρικής Σχέσης, θα πρέπει να έχουν μόνιμο χαρακτήρα. Τι θα γίνει με άλλες φτωχές χώρες, οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται. Όταν μιλάμε για ίση μεταχείριση και δικαιοσύνη σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να έχουν ισχύ οι προσωρινές εμπορικές συμφωνίες. Γι' αυτό υποστηρίζουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πιστεύω ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε ήδη από την πρώτη ανάγνωση. Και το καλύτερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε θα ήταν να φτάσουμε στην τελευταία ανάγνωση στο Συμβούλιο. Η προθεσμία μόνο δεν μας βρίσκει σύμφωνος. Θα πρέπει να την καθορίσουμε και θα ήθελα ο εισηγητής να μας πει κατά πόσο μπορούμε να φτάσουμε σε μια συμφωνία ως προς την ημερομηνία. Ευχαριστώ πολύ. Μια ερώτηση με την μπλε κάρτα για τον κύριο Φιέλνερ από τον κύριο Καμάλ. Πιστείτε, θυμάστε την ερώτηση κύριε Φιέλνερ. Ναι, το περίμενα από σας. Κύριε Καμάλη, του λόγου. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Φιέλνερ που χρησιμοποίησε τον όρο δικαιοσύνη στην ομιλία του. Αν είναι δίκαιο, κατά την άποψή του, να υποχρεωθούν οι χώρες αυτές να μπουν στις διαπραγματεύσεις αυτές και αν είναι δίκαιο να τους στερήσουμε τις ε, προτιμησιακές ε, Μεταχειρήσει επειδή δεν δέχονται να υπογράψουν αυτές τις συμφωνίες οικονομικής εταιρική σχέση, γιατί τι θεωρούν ε, ετεροβαρείς. Κύριος Φιέλνερ, στα αγγλικά. Κοιτάξτε, δεν υποχρεώνει κανεί κανένα να υπογράψει τίποτα. Εμεί έχουμε την δυνατότητα να του δώσουμε την επιλογή αυτή τη διαπραγμάτευση των ΣΟΕΣ. Εάν δεν θέλουν να το πράξουν, θα έχουν τι ίδιε μεταχείρισει με άλλε φτωχέ χώρε. Και δίκαια θα του φερθούμε, ισότιμα δηλαδή, με χώρες εκτός ΑΚΕ. Αλλά το να λέμε ότι επειδή ήταν κάποτε τμήμα, μέρος μιας παράνομης εμπορικής σχέσης, θα πρέπει να συνεχίσουν να έχουν παράνομες εταιρικές προτιμησιακές συνθήκες, ε, δεν νομίζω ότι είναι σωστό και δίκαιο. Ευχαριστώ πολύ και το, κύριο, το λόγο έχει ο κύριος Μπέρντ Λάγκη εκ μέρους των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Στις διαπραγματεύσεις για τις ε, Συμφωνίες Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης έχουμε νομίζω προχωρήσει υπό διαφορετικές συνθήκες Έχουμε μια ευρωπαϊκή, υπό έχουμε μια ευρωπαϊκή επιτροπή με έναν ισχυρό επίτροπο με τους ε, ε, υπαλλήλους, τεχνοκράτες, ειδικού ε, που συζητούν και διαπραγματεύονται με χώρες που έχουν περιορισμένες δυνατότητες. Και έτσι νομίζω θα ήταν και σωστό και εν πάση δεν θα μας κόστησε υπερβολικά να δώσουμε περισσότερο χρόνο και ένα τράτο μεγαλύτερο στις χώρες αυτές. Για να μην δώσουμε και την εντύπωση ότι με την απότομη διακοπή της πρόσβασης στις αγορές αυτές προσπαθούμε να ασκήσουμε πίεση στις χώρες. Βεβαίως και δεν θέλουμε να πιέσουμε κανέναν και να υποχρεώσουμε κανέναν να ε, προσυπογράψει μια ε, οικονομική σχέση που δεν την επιθυμεί. Αλλά θέλουμε να βρούμε λύσεις ε, σε διαπραγμάτευση με τις χώρες αυτές, αποδεκτές και ισότιμες και για τις δύο πλευρές. Μερικές φορές για να το επιτύχουμε αυτό το ε, χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο και γι' αυτό και η σοσιαλδημοκρατική μας ομάδα υποστηρίζει απερίφραστα τις θέσεις του κυρίου Ντέβιτ Μάρτιν, την, ε, παράταση, την ε, χορήγηση δηλαδή, των δύο επιπλέον ετών σε σχέση με την πρώτη επιτροπή, αλλά μόνο των δύο επιπλέον ετών, έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα να βρούμε ένα κοινό πεδίο συνεννόησης. Και παρακαλώ να λάβετε υπόψη το εξή, ότι πρέπει να ακολουθηθεί, πρέπει να γίνει δεκτή αυτή η συμβαστική λύση, την οποία υποστηρίζει η ευρύτατη πλειοψηφία του Κοινοβουλίου και δίνει σαφή μηνύματα, αλλά ταυτόχρονα δεν κλείνει και την πόρτα πραγματεύσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ εκ μέρου των Φιλελευθέρων και Δημοκρατών, ο κύριο Νικολό Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητέ επίτροπε. Υποστηρίζουμε την πρόταση συμβιβασμού στην ίντα. Νομίζω ότι είναι... φτάσαμε σε μια σωστή ισορροπία, έχουμε και μια προθεσμία. Θα ήθελα να λάβετε υπόψη ότι θα ήταν παράλογο να απορρίψουμε την πρόταση της Κομισιόν θα έχουμε δύο χρόνια επιπροσθέτως με βάση και τα αιτήματα που προέρχονται από τις χώρες ΑΚΕ. Νομίζω ότι θα πρέπει να αποδραματοποιήσουμε την κατάσταση γιατί όπως είπε και ο Επίτροπος στην παρέμβασή του μιλάμε για έναν περιορισμένο εμπορικό όγκο όμως σε ορισμένες, για ορισμένες πρωτεύουσες των χωρών ΑΚΕ η αυριανή απόφαση έχει μεγάλη σημασία διότι υπάρχει μεγάλη ασυμμετρία μεταξύ διακυβεύματος και ορισμένων χωρών και δεν νομίζω ότι με μία τόσο κοντινή προθεσμία θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε μία ταχεία ε, έκβαση των διαπραγματεύσεων. Εμείς θέλουμε τις ΣΟΕΣ αυτές είναι όμως εταιρικέ συμφωνίες. Θα πρέπει να φτάσουμε σε αυτές με την πυθό, με τη δύναμη της πυθούς. Γι' αυτό νομίζω ότι μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια, τα επιπρόσθετα δύο χρόνια, θα μπορέσουμε να καταβάλουμε μεγαλύτερες προσπάθειες διαπραγμάτευσης, διευρύνοντας και το δίκτυο συνομιλητών μέσα στα πλαίσια και της κοινωνίας των πολιτών αυτών των χωρών, να έρθουμε σε επαφή με τα εθνικά κοινοβούλια. Πολλές φορές δεν κυρώνουν, όμως έχουν πολιτική φωνή μέσα στα πλαίσια των εθνικών ε, συζητήσεων και πολλές φορές παραπονούνται ότι δεν λαμβάνουν επαρκείς πληροφορίες. Ίσως θα πρέπει να προωθήσουμε και σεμινάρια στις χώρες ε, ΑΚΕ με τη συνεργασία της ΜΚΙΟ οι Κενιάτες λένε θέλουμε να πάμε ε, μακριά, ας πάμε μακριά από κοινού. Εξ ονόματος των Πρασί, η κυρία Κέλλερ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ με την πρόταση να αποκλειστούν από, τις, ε, από την προτιμησιακή πρόσβαση στι αγορέ τα αναπτυσσόμενα κράτη. Προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τα πιέσει, να προσπογράψουν ε, εμπορικέ σχέσει. Δεν πρόκειται για τα συμφέροντα των κρατών αυτών, αλλά για τα συμφέροντα μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι για την, ανάπτυξη των κρατών, των εταίρων. Κράτη όπως το Καμερούν, η Ακτή του Ελεφαντοστού, η Ναμίμπια κινδυνεύουν να υποστούν βαρύτατο πλήγμα από τον αποκλεισμό αυτό και εάν η Κένια προσπογράψει μια συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης θα χάσει ε, σημαντικές οικονομικές δυνατότητες. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι προσπαθούμε να υποχρεώσουμε τα κράτη αυτά να αγοράζουν τα δικά μας εμπορεύματα και μόνο. Αλλά αν θέλουμε πραγματικά την ανάπτυξη των αυτών, δεν θα πρέπει να τα εμποδίζουμε να επιλέγουν μόνο τους τις εταιρικές σχέσεις που θέλουν να συνάψουν. Σας ευχαριστώ εκ μέρους της Ενωτικής Αριστεράς, ο κύριος Σόλτς. Κύριε Επίτροπε Ντεγκούχτ, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, συζητούμε σήμερα μια πρόταση δική σας κύριε Επίτροπε, η οποία νομίζω επιφέρει, μπορεί να επιφέρει βαρύτατο πλήγμα στο κύρος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε εταίρους στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων που εσείς θέλετε να πιέσετε και να εκβιάσετε να συνάψουν συμφωνίε οικονομική εταιρική σχέση. Έτσι λοιπόν χάνεται κάθε αξιοπιστία και κύρος Ευρωπαϊκής Ένωσης ως δίκαιου παράγοντα ε, και εταίρου στις ε, διεθνείς εμπορικές σχέσεις. Η Επιτροπή Ανάπτυξης έχει γνώσεις και ιδιαίτερη ευαισθησία έναντι των κρατών αυτών ε, της ε, Αφρικής, καραβικής και του Ειρηνικού και έχει απορρίψει και μέσω της ε, Προέδρου του και Προέδρου της ομάδας μου, κυρίας Γκαμπιτσίμερ, Όλε αυτέ τι προτάσει τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καλό, λοιπόν και όλου του συναδέλφου, εκ μέρου τη ομάδα μου, αγαπητοί συναδέλφοι, κυρίω εσεί της Επιτροπής ε, ανάπτυξη, να απορρίψετε αυτές τις τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μην ανατρέψετε μέσα σε μια βραχυπρόθεσμη και μια κοντόφθαρμη προσέγγιση τι δεκαετίες αυτές αναπτυξιακή συνεργασία. Κύριε Επίτροπε, κύριε Ντεγκούχτ, έχει δυναμικό εκρηκτικό για, τις, ε, για τη συνεργασία με τι χώρε Αφρική η πρόταση κινδυνεύει να απομονωθεί και σε σχέση με τις χώρες γειτονίας της ε, και να χαθεί και η ευκαιρία για καλή αναπτυξιακή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσείς ε, κατηγορείτε άδικα τους ε, ε, Αφρικανούς και προσπαθείτε να τους τιμωρήσετε για καθυστερήσεις για τις οποίες είστε εσείς οι ίδιοι υπέτεια. υπέτειοι. Γιατί πρέπει να καταργηθούν ε, οι εξαγωγικοί δασμοί που επιβάλλουν τα κράτη αυτά. Μόνο στις πρώτες σύλλες στο προϊόν της εξορρυκτικής της βιομηχανίας επιβάλλει να μπει παραδείγμα τέτοιου είδους εξαγωγικούς δασμούς. Είναι δυνατόν να τους απαγορεύσουμε κάτι τέτοιο. Πρέπει λοιπόν ε, να αναγνωριστεί ότι αυτές οι προτάσεις της Επιτροπής, Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι απολύτω αντίθετε με του αναπτυξιακού στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σας καλώ να την, να την αποσύρετε την πρόταση αυτή. Ευχαριστώ ο Πρόεδρος και τώρα οι λοιποί ομιλητές. Ο κύριο Βιντάλ Μορέιρα πρώτο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτή η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γύρει δύο ερωτήματα. Θα πρέπει να αρθούν τα μονομερή προτιμησιακά μέτρα προς χώρες ΑΚΕ και ε, σε ποιες χώρες θα πρέπει να ισχύει και ποιο, καθεσ, καθεστώς θα πρέπει να ισχύει για τις χώρες που δεν εντάσσονται στο, στις χώρες ΑΚΕ και συμφωνίες Κοτονού. Επίσης, ε, τι θα γίνει όταν ε, δεν υπάρχει προθεσμία, διότι παλαιότερα δυστυχώς δεν υπήρχε προθεσμία. Πιστεύω ότι ο κανονισμός του 2007 ήταν μεταβατικός και νομίζω ότι μέσα στα πλαίσια των γενικευμένων προτιμήσεων εκρίθη ότι οι γενικευμένες αυτές προτιμήσεις ήταν παράνομες σύμφωνα με τον ΠΟΕ. Θα πρέπει να δούμε κατά πόσο λοιπόν αυτές οι μονομερείς εμπορικές προτιμήσεις θα τις εντάξουμε στις χώρες ΑΚΕ και ιδιαίτερα για τις χώρες που δεν την χάνουν αυτού του καθεστώτος μέσα στα πλαίσια της ε, συμμετοχής αυτής διαδικασίας. Ως προς την προθεσμία, η ίντα δεν έχει πιστεί από τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γι' αυτό ζήτησε παράταση της προθεσμίας κατά δύο έτη, δηλαδή μέχρι το 2000, από το 2014 στην 1η Πρώτου 16. Είναι πιο ε, σωστή αυτή η προσέγγιση και μπορούμε έτσι να διευρύνουμε αυτή την προθεσμία χωρίς να παρατείνουμε ε, υπερβολικά αυτό το παράνομο καθεστώς των εμπορικών συμφωνιών που ήδη ισχύουν. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μέρφυ για ένα λεπτό. Νομίζω ότι η πρόταση αυτή για την κατάργηση των ρυθμίσεων των αφορολογήτων ουσιαστικά έχει ένα όνομα, εκβιασμός. Αυτό θα κλείσει την ευρωπαϊκή αγορά για ορισμένους τομείς και θα είναι κάτι το καταστροφικό για τις χώρες αυτές. Για την Αμίμπια, σαν παράδειγμα, οι δεσμοί που θα ζητηθούν και θα επιβληθούν για ε, το βοηθοί θα τους κάνουν να χάσουν το 60% του κέρδους από τις εξαγωγές τους. Εμείς πρέπει να αυξήσουμε τις πιέσεις βέβαια προς τις χώρες αυτές για να υπογράψουν τις συμφωνίες στην ΕΠΑ, Ξέρετε ότι έχουν υπάρξει πάρα πολλές διαφωνίες γύρω από τις συμφωνίες αυτές σε αυτές τις χώρες και δεν θα πρέπει να τις πιέσουμε με απαράδεκτους τρόπους γιατί βλάπτουμε όχι μόνο τις οικονομίες γενικότερα των χωρών αυτών, αλλά τους φτωχούς αγρότες κυρίως. Και έτσι λοιπόν η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να απορριφθεί. Η κυρία Μπαντία Ικουτσέτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, Αναρωτηθήκατε γιατί πρέπει να δώσουμε περισσότερο χρόνο σε ορισμένες χώρες ε, μέσα στα πλαίσια των συμβάσεων για τις χώρες ΑΚΕ. Νομίζω ότι δεν είναι έτοιμοι όλοι για κάτι τέτοιο, διότι μιλάμε για δυσχερείς οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες. Θέλουμε να προχωρήσουμε με αυτές τις χώρες, θέλουμε να προχωρήσουν ή τις αφήνουμε σε μια επισφαλή θέση την οποία κατέχουν τώρα. Γι' αυτό πιστεύω ότι η ημερομηνία του 2016 που προτείνουμε θα επέτρεπε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και θα δίναμε και μεγαλύτερη νομική ασφάλεια στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και σε αυτές τις χώρες οι οποίες θα πρέπει να προωθήσουν την ανάπτυξή τους. Νομίζω ότι αυτή η επέκταση των δύο χρόνων δεν σημαίνει ότι παραβαίνουμε τα πλαίσια λειτουργίας που μας έχει θέσει ο ΠΟΕ. Γι' αυτό θα ζητήσω την παράταση, την διετή παράταση και ελπίζω να ληφθεί υπόψη. Ο κύριος Κάσμαν. Ευχαριστώ. Ανησυχώ γιατί πιστεύω ότι οι χώρες ΑΚΕ και οι κυβερνήσεις τους υφίστανται πιέσεις για να υπογράψουν τις ΣΟΕΣ χωρίς να γνωρίζουν επακριβώ τους όρου. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν αυτές οι χώρε. Μιλάμε για την περιφερειακή ολοκλήρωσή του και η Ευρώπη ξέρει ότι κάτι τέτοιο χρειάζεται χρόνο. Επειδή έχω ασχοληθεί με τις σχέσεις μας με την Νότιο Αφρική, νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ε, συγκεκριμένες συνθήκες έτσι ώστε να ισχύσουν οι ΣΟΕΣ. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτή η προθεσμία θα μπορούσε να σταθεί γκυγιωτίνα και να μην βοηθήσει αυτές τις χώρες. Γι' αυτό, όπως είπε και ο συνάδελφός μας, ο, ο Μάρτιν θα μπορέσουμε να παρατείνουμε αυτή την προθεσμία μέχρι το 2016 έτσι ώστε να δούμε πώς θα ορίσουμε και το νέο γύρο, τη νέα συμφωνία Κοτονού, γιατί αυτή τη φορά δεν έχουμε περιθώρια ασφάλματος. Τώρα αρχίζουμε με τη διαδικασία Catch the Eye. Ο κύριος Ζουάου Φερέιρα ζήτησε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αυτή η πρόταση κανονισμού αποτελεί εκφοβισμό και εκβιασμό μέσα στα πλαίσια των οικονομικών εταιρικών σχέσεων με τις χώρες ΑΚΕ. Δηλαδή επικρατεί το διέρη και βασίλευε. Αυτή είναι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δηλαδή πιέζετε τις χώρες έτσι ώστε στη συνέχεια να μπορέσετε να δρέψετε τους καρπούς. Αυτό θα ήταν ολέθριο για τις χώρες ΑΚΕ και γι' αυτό ανθίστανται πολλές από αυτές πολύ σωστά ανθίστανται και θα πρέπει να μην υποκύψουν στις πιέσεις. Επίσης θα πρέπει να προωθήσουμε τις ε, συμφωνίες συνεργασίας μέσα στα πλαίσια της εθνικής κυριαρχίας τους, χωρίς να μιλάμε για νέο απικισμό ε, υποσκάπτοντας την εθνική κυριαρχία αυτών των χωρών. Ο δεύτερος ο ομιλητής είναι ο κύριος Τυρολίων. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όλοι γνωρίζουμε πόσο οι διαπραγματεύσεις για τις συμφωνίες αυτές είναι χρονοβόρες και δύσκολες και γι' αυτό και εγώ έχω δύο απόψεις να πω γύρω από το ένα θέμα, από το συγκεκριμένο θέμα. Βλέπουμε ότι μόνο 18 από τις 36 χώρες που έχουν υπογράψει τις συμφωνίες αυτές τις έχουν επικυρώσει. Οι άλλες καλούνται να το κάνουν αυτό το ταχύτερο δυνατόν γιατί αλλιώς οι προσπάθειές τους θα καταστραφούν το 2014. Από την άλλη γνωρίζαμε ήδη από το 2007 ότι ο κανονισμός αυτός δεν θα ήταν παρά προσωρινός και ασύμβατος με τους κανόνες του ΠΟΕ. Συνεπώς, η πρόταση του εισηγητή μας είναι η καλύτερη συμβιβαστική λύση έτσι ώστε οι υπηρεσίες της Επιτροπής και οι χώρες ΑΚΕ να έχουν τον απαιτούμενο χρόνο για να κλείσουν τις διαπραγματεύσεις έγκαιρα. Αν αύριο δεν υπάρξει πλειοψηφία στην ψηφοφορία για το 16, τότε θα ζητήσω από τους συναδέλφους να απορρίψουν την πρόταση της Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Θα μπορούσα να ζητήσω και εγώ το λόγο, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ. Θα ήθελα. Θα ζητήσω από τον Επίτροπο να κλείσει τώρα τη συζήτηση. Κύριε Ντεχούχτ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αν θέλετε να σας δώσω ένα χρόνο από τον χρόνο που έχω στη διάθεσή μου. Εκτός ε, βέβαια αν θέλετε να με διακόψετε μετά για υπέρβαση. Κατανοώ πολλές από τις παρατηρήσεις οι οποίες έγιναν και γι' αυτό θα ήθελα να σας ζητήσω να μείνουμε στα γεγονότα. Αυτό για το οποίο πρόκειται είναι ότι ορισμένες χώρες δεν έχουν ακόμα υπογράψει ή επικυρώσει μια συμφωνία η οποία ολοκληρώθηκε το 2007. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μιλάμε για το τι έγινε στο παρελθόν δηλαδή, σαφώς. Το ότι θέλουμε εμείς να υποχρεώσουμε τις χώρες αυτές να κλείσουν, να εγκρίνουν και να επικυρώσουν ε, τέτοιου είδους συμφωνίες, τις συμφωνίες ΕΠΑ, δεν είναι κάτι το οποίο στέκει. Εγώ αναφέρθηκα σε οκτώ χώρες, οκτώ χώρες οι οποίες με τον ένα ή άλλο τρόπο επηρεάζονται από τις προτάσεις μας. Θα τις ξαναπώ τις χώρες αυτές. Καμερούν, Ακτή Ελεφαντοστού, Φίτζι, Γκάνα, Κένια, Σουαζιλάνδη. Πρόκειται για χώρες χαμηλών εισοδημάτων και δύο, Μποτσουάνα και Ναμίντια, οι οποίες είναι μεσαίες προς τα άνω χώρες. Δεν ε, καταλαβαίνω λοιπόν γιατί πιστεύετε ότι εμείς θα φίξουμε τις αναπτυσσόμενες χώρες. Τις αναπτυσσόμενες χώρες έχετε δύο διαφορετικές κατηγορίες. Έχετε τις LDCs που έχουν ε, τις χαμηλότερο επίπεδο, που έχουν ε, ωφεληθεί στο παρελθόν και έχετε και τις ανωτέρω επίπεδου οι οποίες έχουν επωφεληθεί πολύ από τις συμπληρωματικέ συμφωνίες GSP και GSP+. Λοιπόν, εμείς λέμε στις χώρες αυτές ότι αν δεν προχωρήσετε στην εφαρμογή αυτών των ρυθμίσεων ε, πάντα είχαμε πει ότι από όλη αυτή τη μεγάλη κατηγορία των χωρών κάποιες χώρες θα μείνουν με μονομερείς μορφές πρόσβασης στις ευρωπαϊκές αγορές έτσι ώστε να μπορούν να εξάγουν τα προϊόντα τους χωρίς ποσοστώσεις και να εξάγουν τα προϊόντα τους χωρίς δασμούς. Δεν δημιουργούμε λοιπόν εμείς καμία μορφή ανισότητας ανάμεσα στις 6 ή 8 από τη μία χώρες και στις 60 χώρες από την άλλη. Δεύτερον, Υποχρεώνουμε κάποια από τις χώρες αυτές να το κάνει αυτό. Όχι βέβαια, αν δεν θέλουν να εγκρίνουν την συμφωνία την οποία οι ίδιες συνήψαν το 2007, μπορεί και να μην το κάνουν. Και πάντα εμείς θα συνεχίσουμε να διαπραγματευόμεθα μαζί τους. Αλλά δεν βλέπω γιατί εμείς θα ήμασταν άδικοι, πιεστικοί, βίαιοι, εκβιαστές όταν ζητάμε από κάποιον ο οποίος υπέγραψε μια συμφωνία πριν πέντε χρόνια, μια συμφωνία που είχε γίνει αντικείμενο διαπραγμάτευσης τρία-τέσσερα χρόνια και έπρεπε να ξεκινήσουν οι αλλαγές ήδη εδώ και δώδεκα χρόνια βέβαια, Εσείς υποσχεθήκατε ότι θα το επικυρώσουν. Είχατε πέντε χρόνια στη διάθεσή σας ή εφτά χρόνια, εξαρτάται πότε ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις. Και εμείς δίνουμε μισή χρόνο ακόμα για να επικυρώσετε, όχι να διαπραγματευτείτε μια νέα συμφωνία. Λοιπόν, αυτό είναι εκβιασμός, αυτό είναι βίαιη πίεση. Δεν το πιστεύω εγώ αυτό. Ο Μπεν Λάγκε είπε ότι Υπάρχει αντιπαράθεση ανάμεσα σε μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε ασθενείς χώρες. Ευχαριστούμε καταρχάς που μας ονομάζεται ισχυρό όργανο. Αλλά ξέρετε ότι οι χώρες αυτές, κάποιες από αυτές είναι ασθενείς, αλλά δεν αναφέρομαι στις ασθενέστερες των χωρών αυτών. Αναφέρομαι σε χώρες οι οποίες είναι αρκετά αναπτυγμένες. Δεν αναφέρομαι εγώ στις κατωτέρου οικονομικού εισοδήματος χώρες. Το θέμα δεν είναι αν οι χώρες αυτές είναι ισχυρές ή αδύναμες. Το θέμα είναι εάν πράγματι επικυρώσουν αυτό το οποίο έχουν συμφωνήσει στο παρελθόν. Αν αναλάβουν δηλαδή τις υποχρεώσεις τις οποίες είχαν αναλάβει εδώ και αρκετό καιρό. Και μια τελευταία παρατήρηση. Πράγματι το εμπόριο μπορεί, ε, είπατε ότι μπορεί να, να προωθήσει την ανάπτυξη. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Βλέπετε ότι με τα υπάρχοντα προγράμματα ο όγκος των εμπορικών συναλλαγών κατεβαίνει δραστικά. Γιατί? Γιατί το εμπόριο δεν είναι το να εξάγει κανείς κάποια προϊόντα σε άλλη αγορά. Είναι να εμπλακεί με την αγορά αυτή, να έρθει σε σχέση με την αγορά αυτή να υπάρξουν εμπορικές συναλλαγές και προς τις δύο κατευθύνσεις. Το εμπόριο επιτρέπει να δημιουργηθεί ένα εμπορικό πλαίσιο θα έλεγα μέσα στο οποίο θα γίνουν περισσότερα πράγματα από ό,τι στο παρελθόν. Λυπάμαι γιατί οι εμπορικές συναλλαγές μας με την Αφρική μειώνονται. Θα έπρεπε να αυξάνονται. Λυπάμαι γι' αυτό. Θα ήθελα να είμαι πολύ ευέλικτο σε σχέση με τις συμφωνίες ΕΙΠΑ, τις οποίες πρέπει να διαπραγματευτούμε ακόμα. Με την ασυμμετρία εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, καμία προκατάληψη. Ας μπορέσουν οι χώρες αυτές ε, να εξάγουν περισσότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με νέες εμπορικές ρυθμίσεις, με νέες διευκολύνσεις. Συμφωνούν και οι συνάδελφοί μου με αυτό αλλά παρόλα αυτά πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να αναγνωρίσουν τις ανηλυμένες τους υποχρεώσεις έτσι ώστε το νομικό σύστημα και τα νομικά δικαιώματα τα οποία προέρχονται από το διαπραγματευμένο πλαίσιο να είναι σε ισχύ. Γι' αυτό λοιπόν ακριβώς και εμένω με την πρόταση την οποία σας έκανα και ελπίζω ότι αύριο όταν ψηφίσετε θα το λάβετε υπόψη σας. Δεν είναι η πρότασή μας κατά των αναπτυσσομένων χωρών, δεν είναι η πρότασή μας κατά της Αφρικής, είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει να οριμάσουν οι εμπορικές μας σχέσεις με ορισμένες χώρες οι οποίες πρέπει να αναπτυχθούν ακόμα. Οι χώρες που δεν έχουν απογειωθεί ακόμα οικονομικά είναι οι χώρες της υποσαχαρικής Αφρικής. Αυτό δεν γίνεται τυχαία, είναι καθήκον μας λοιπόν κάτι να κάνουμε γύρω από αυτό. Ευχαριστώ Επίτροπε. Ο κύριος Μάρτιν τις τελικές του παρατηρήσεις. Κύριε Επίτροπε, πρέπει να εξηγήσετε στο σώμα γιατί ορισμένες χώρες που έχουν υπογράψει τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης και ακόμη δεν τις έχουν κυρώσει. Και το σήμερα και ο κύριος Κάσμαν και άλλοι συναδελφοί ότι αυτές οι συμφωνίες έχουν σαν στόχο κυρίως την περιφερειακή ολοκληρώση. Έχουμε λοιπόν θέσει ορισμένες από τις χώρες αυτές, αν όχι σε αδύνατη, πάντως σε πολύ δύσκολη θέση. Και ε, σαν παράδειγμα, σας φέρνω την ε, Κένια, η οποία εάν προσυπογράψει, εάν κυρώσει μάλλον μονομερός την ε, Συμφωνία Οικονομική Εταιρική σχέση, διαρριγνεί του δεσμούς τη με, την Ανατολική, με τις χώρες Ανατολικής εάν δεν το πράξει και δεν κυρώσει, έχει οικονομική ζημιά. Θα αντιμετωπίσει πολύ υψηλού δασμούς εάν περάσει αυτή η πρότασή σας και δεν έχει κυρώσει ακόμη την ΣΟΕΣ Κένια και ταυτόχρονα η Επιτροπή και το Κοινογύλιο φαντάζομαι θα ε, συμφωνήσει σε μια ε, σχέση εταιρική οικονομικής σχέσης με την Κολομβία, ένα από τους κύριους ανταγωνιστές για τα προϊόντα τους, ε, της Κένιας, στην οποία θα δώσει προτισμιακές ε, σχέσεις. Άρα λοιπόν αυτό που λέω είναι μόνο ένα τράτο δύο ετών για να μπορέσουν και τις σχέσεις με τους εταίρους από την Ανατολική Αφρική και την ΣΟΕΣ να ακυρώσουν οι Κενιάτε. Αλλά το ίδιο ισχύει όχι μόνο για την Κένια, μια και δεν έχω χρόνο, δεν μπορώ να αναπτύξω περισσότερα τα επιχειρήματα για την Αμίμπια, για την ε, Νότια Αφρική και για άλλε χώρε. Εσεί λέτε το 2014, κύριε Επίτροπε, γιατί λέτε ότι έτσι έχουν περισσότερη δύναμη και πιεστική ε, πυθό οι διαπραγματεύσει. Εγώ όμω γι' αυτόν ακριβώ το λόγο δεν θέλω το 2014 ω προθεσμία, γιατί είναι πολύ, πιεστικός ακριβώς, ε, πολύ πιεστική ακριβώ αυτή η προθεσμία και γιατί δεν είναι έτοιμε οι χώρε. Και όπω είπα, α μην βιαζόμαστε, α μην πιέζουμε και α ορίσουμε μια προθεσμία συγκεκριμένη, όχι ευέλικτη, όχι μεταβλητή. Άπαξ και περάσει η νομοθεσία αυτή, το νομοθέτημα αυτό, θα ισχύει το 2016 και θα έχουν χρόνο οι χώρες αυτές της Αφρικής να προσαρμοστούν ταυτόχρονα όμω και εμεί από πλευρά μα θα δείξουμε περισσότερη λογική κοινή λογική και ευελιξία. Ευχαριστώ πολύ. Κλείνει εδώ η συζήτηση. Προφορία αύριο στι 12. Σας ευχαριστώ. Και περνούμε τώρα στο προσεχές θέμα της ημερησία διάταξη. Που είναι η έκθεση του κύριου Κάρενς. Διακυβερνητικές συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών στον τομέα της ενέργειας.